οι οποίες προκαλούνται από τον άνθρωπο και εγώ ήμουν και σκιώδης εισηγήτρια στην έκθεση αυτή. Ε, τα ψηφίσματα αυτά δυστυχώς ε, πολύ δύσκολα μεταφράζονται στην πράξη και δεν είναι και πολύ αποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται. Θα πρέπει λοιπόν το ζήτημα να ξανασυζητηθεί ε, και κάθε φορά θα, αν δεν το λύσουμε θα βρισκόμαστε εδώ να το συζητάμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις μονόλεπτες παρεμβάσεις. Στο επόμενο σημείο έχουμε την ολοκλήρωση εσωτερική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου από τον κύριο Πάμπλο Αρία Ετσεβέιρα. Είναι η έκθεση. Έχετε το λόγο, κύριε Σιγητά, για τέσσερα λεπτά. Καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζετε όλοι, το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες σημαίνουν ότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την οικονομία μας σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ε, έχουμε καθημερινά. Οι νέε τεχνολογίε μέσω διαδικτύου που έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε δεν υπήρχαν πριν από κάποια χρόνια. Πλέον όμως είναι γεγονός και πολύ σύντομα θα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη τη καθημερινή μας ε, ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να, βρεσκούμε, να βρεθούμε στο ύψο των περιστάσεων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες ε, για τους πολίτες που θα επιλύσουν ε, τα σημερινά προβλήματα και θα προσαρμοστούν στο αύριο. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να αναλάβουμε ω ευθύνη προκειμένου να ε, προετοιμάσουμε το έδαφος για αυτά τα οποία ε, περιμένουμε στο μέλλον. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους φραγμούς που σήμερα αποτελούν πρόσκαιωμα προς αυτό το σκοπό. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα όπλο στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, καθώς επίσης και να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για ένα όπλο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αξία και να δημιουργήσει και πάρα πολλέ δυνατότητε και για του πολίτε αλλά και για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, ειδικά σε περίοδο κρίση. Γι' αυτό λοιπόν οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αρθούν οι υπάρχοντε φραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη και να εμπιστευτούμε αυτό το μέσο, να το απλουστεύσουμε και να του προσδώσουμε τη δέωσα διαφάνεια ε, κυρίως ως προς τους κανόνες που το διέπουν. Έτσι θα μπορέσουν οι πολίτες να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες δυνατότητε που προσφέρει. Μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια αγορά και θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και να δείξουμε το δέον ηγετικό ρόλο, αλλιώς θα, θα βρεθούμε ε, στα μετόπιστε και θα πρέπει να μπορέσουμε να προάγουμε το διαμεθοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε όχι μόνο την εσωτερική αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά να συμπληρώσουμε την, ε, ε, το εσωτερικό εμπόριο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία προτείνω θέλω να βελτιώσουν την πρόσβαση ε, στο διαδίκτυο στην Ευρώπη, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στους καταναλωτές μέσω ενός ευρωπαϊκού σήματος και να ενισχύσουν την εποπτεία και την επιτήρηση του δικτύου και να δημιουργήσουν δημιουργήσουν ενημερωτικές εκστρατείε, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν πώς να ε, διαμαρτυρηθούν εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχουν προβλήματα. Επίσης, ε, μας ενδιαφέρει η προστασία της ιδιωτικής ζωή και των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στου επιχειρηματίες να πολλούν τα προϊόντα τους ε, online, διευκολύνοντας τις πληρωμές και υιοθετώντα και μέτρα για τη φορολογία αν χρειαστεί απαραίτητο. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία του να προστατεύουμε τους ανηλίκους ε, στη χρήση του διαδικτύου. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να ενισχύσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και για να ε, έχουμε ε, κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν και για το μέλλον, το οποίο ζούμε ήδη. Θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών μας και θα ενισχύσουν τις οικονομίες μας και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίς φραγμούς. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω εδώ την υποστήριξή σας για να προχωρήσουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, ευχαριστώ. Τώρα θα αρχίσουμε τη διαδικασία Catch the Eye θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε 11. Έχω ε, πέντε ομιλητές, την κυρία Ρόντοβα, Κιτάου, ο Πάσκα, Έλλη. Λυπάμαι για τους υπολείπους. Μπορείτε όμως να υποβάλλετε δηλώσεις γραπτός σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Ρόιτοβα. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι διαπιστώνω ότι ο εισηγητής ε, βασίστηκε στην έκθεσή μου σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταλανοτών που είχε υιοθετηθεί στην προηγούμενη θητεία. Και παρόλο που έχει αυξηθεί πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο, ακόμη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι δυνατότητες ε, και δεν έχουμε προσελκύσει τους πελάτες από άλλες ε, χώρες μέλη. Ε, ε, γίνεται μία τεχνητή διαχείριση των τιμών παρόλο που υπάρχουν δυνατότητες. Χαίρομαι λοιπόν διότι ο εισηγητής προσπαθεί να βελτιώσει τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου επισημένοντας όμως ε, και τις παγίδες, την πορνογραφία, την ε, διακίνηση παρανόμων ε, εμπορευμάτων και την προστασία των παιδιών που ελπίζω ότι θα προστατευτούν καλύτερα από, τα, από την Επιτροπή, από τους παρελθόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. βλέπουμε ότι αυξάνονται οι δυνατότητες που προσφέρονται στον καταναλωτή για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αγορά. Ε, στηρίζουμε τις ε, δυνατότητες οι οποίες δίνονται ε, διευρωπαϊκά για να υπάρξει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε σύντομα μία αρχή η οποία θα εποπτεύει τις ηλεκτρονικές υπογραφές και συγχρόνως ζητήσουμε ζητούμε από την Επιτροπή ε, να ε, αναλάβει την πρωτοβουλία για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2020 και τουλάχιστον ελπίζω μέχρι το 2015 το ίμις των ε, δημοσίων αγορών θα γίνεται ηλεκτρονικά όπως αποφασίστηκε στο Μάντριστερ το 2005 στο συνέδριο e-government. Η κυρία Φιγκερέντο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω τρία θέματα που μου φαίνονται σημαντικά σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν διευκρινήσεις στα θέματα αυτά. Καταρχήν θα πρέπει να συμβιβάσει κανείς τα δικαιώματα του καταναλωτού και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα του παιδιού και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών ούτε να τα διακινδυνεύσουμε και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι στόχοι οι οποίοι έχουν όμως ε, καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρική σχετικά με την ευρυζώνια ε, χρήση θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί μέχρι το 2013 και ξέρουμε ότι περίπου 30% των οικογενειών δεν δεν έχουν καν τη δυνατότητα για μία απλή σύνδεση με το διαδίκτυο. Οπότε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει αυτή την ευρυζώνια χρήση σε όλα τα άτομα ε, μέχρι την ημερομηνία του 2013. Ο κύριος Πασκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ηλεκτρονικών πωλήσεων, αλλά υπάρχουν πολλές κουλτούρες σε πολλές χώρες. Σε διάφορες χώρες μερικά φαρμακευτικά ε, προϊόντα, προϊόντα πολλούνται χωρίς συνταγή, ενώ σε άλλες χώρες χρειάζονται συνταγή. Ε, ε, υφίστανται ρυθμίσεις. Αλλού πολλούνται εύκολα πορνογραφικά προϊόντα, ενώ σε άλλες χώρες δεν πολλούνται καθόλου το να ανοίξουμε την ηλεκτρονική αγορά θα πρέπει ε, να προστατεύσουμε αυτούς τους κανόνες, αυτές τις κουλτούρες τις χώρες ε, όπου ε, πάρα πολλοί σκέφτονται ότι πρέπει να προστατευθούν οι νέοι και τα παιδιά το ηλεκτρονικό εμπόριο ευεργέτησε τόσο τις επιχειρήσεις όσο τους καταναλωτές. Υπάρχει επίσης όμως μια άποψη που δεν με ικανοποιεί, είναι το e-ticketing δηλαδή τα εισιτήρια τα που πολλούνται ηλεκτρονικά για αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πολλούνται σε τρομερές τιμές, πράγμα που δεν πρέπει να είναι αποδεκτό. Έχουμε 70 ε, ευρώ πολλούνται ε, εισιτήρια για ποδεσφορικούς αγώνες από έναν οργανισμό. Ε, εάν Ήτανε καρτέλ θα συλλαμβάνονται, αλλά στο διαδίκτυο ε, πολλούνται ακόμα και με 500 ευρώ. Ε, βεβαίως πολλούν εισιτήρια επειδή υπάρχει ζήτηση. Είναι μια πρακτική αθέμητος ε, και νομίζω ότι υποβαθμίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα πρέπει να είναι προς όφελος των καταναλωτών. Ο κύριος Ντεγκούχτα για την Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Αρία Σετσεβερία, τον εισηγητή, το κοινοβούλιο ολόκληρο ε, για αυτήν την ευρία αξιολόγηση της ηλεκτρονικής αγοράς. Νομίζω ότι εν ευθέτω χρόνο ήρθε αυτή η εισήγηση και μας υπενθυμίζει ότι για πάρα πολλές επιχειρήσεις και καταναλωτές η ηλεκτρονική αγορά δεν είναι πραγματικότητα, διότι λείπουν ορισμένοι κρίκη στην εσωτερική αγορά. Οι πολλοί καταναλωτές γνωρίζουν ε, την εσωτερική αγορά αγοράζοντας ηλεκτρονικά διαμέσω του ε, διαδικτύου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να αναπτύξουν νέες αγορές ε, διαμέσου του διαδικτύου. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές ούτως ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά που να γίνει πραγματικότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε τα κενά στην εσωτερική αγορά και για να αποδώσει καλύτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει η Κομισιό να δει ποια θα είναι αντίδραση σε αυτήν την έκθεση. Πάρα πολλά από αυτά τα σημεία έχουν, εξετάζονται στην ψηφιακή ατζέντα. Η έκθεση δείχνει δύο οδούς που θα πρέπει να διερευνήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διευκολύνουμε την ζωή ζωή και να την κάνουμε πιο απλή για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές εναρμονίζοντας κανόνες παραδείγματος χάρη και διαδικασίες ε, για να είναι λιγότερο δαπανηρή η διαδικασία για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές, ε, τα θέματα ε, δικαιωμάτων, τα τιμολόγησης κλπ. Η Επιτροπή υποστηρίζει μια οδηγία ε, σχετικά με τους καταναλωτές που εξετάζεται και τώρα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Θα διευκολύνουμε τη ζωή των καταναλωτών με καλύτερη νομοθεσία, κυρίως με την οδηγία υπηρεσιών που απαγορεύει τις γεωγραφικές διακρίσεις κατά των καταναλωτών σε σχέση με τις παραδόσεις και την πληρωμή. Επίσης είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου για να μπορέσουν ε, επίσης ε, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να έχουν επαφές με την γραφειοκρατία, με απλούστερες διαδικασίες ε, που θα έχουν μόνο μία στάση στην όλη διαδικασία, μία μόνο θηρίδα. Επίσης, ε, θέλουμε να βρούμε λύσεις εξετάζοντας δυνατότητες να μπορεί να υπάρξει ένας κώδικας ε, για διαδικτυακά δικαιώματα. Θα πρέπει ε, να εφαρμόσουμε καλύτερα τους κανόνες, να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Επίσης, επίλυση των διαφορών με χαμηλό κόστος, ταχύρυθμη διαδικασία που θα διευκολύνει τις αγορές ε, στο διαδίκτυο από τους καταναλωτές. Θα πρέπει να έχουμε μια πρόταση για ένα σύστημα διευθέτησης των διαφθορών μέχρι το 2012. Επίσης έχουμε την πρόθεση να εξασφαλίσουμε οι καταναλωτές σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μαζικές διεκδικήσεις θα μπορούν να λάβουν αποζημιώσεις και επανορθώσεις για επίσης προτάσεις για συλλογική επανόρθωση για το 2011 γνωρίζοντας ότι οι δημόσιες αρχές ε, παρακολουθούν την εσωτερική αγορά ως θεμέλιο για να υπάρξει εμπιστοσύνη. Η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών ε, και οι Εθνικές Αρχές προσπαθούν να καταπολεμήσουν αθέμητες πρακτικές στο διαδίκτυο. Επίσης, εμείς παρακολουθούμε Επίσης το, το scoreboard όπου γίνεται βαθμολόγηση των διαφόρων περιπτώσεων. Στην αρχή του 2011 μια ανακοίνωση θα αφιερωθεί στην αξιολόγηση α, της εφαρμογής της οδηγίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιείται καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά όσους ασχολήθηκαν με αυτήν την έκθεση η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και λυπούμε που ο κύριος Ντάλι είναι απόν για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ετσεβερία για την έκθεσή του και αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Ε, το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της κυρίας Γκάλλο.